Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανθρωπιστική και πολιτική κρίση που υπάρχει στην Ουγγαρία. Θα ήθελα να υποβάλω μία πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στη διάσκεψη των Προέδρων. Δηλαδή, να μεταβούν αυτοκίνητα ε, του Κοινοβουλίου προς την Ουγγαρία για να λάβουν ορισμένους ετούντες άσυλο και πρόσφυγες και να τους υποστηρίξει. Αυτό θα ήταν και μια συμβολική κίνηση και δείχνει τη θέση μας έναντι της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ για αυτήν την υπόδειξη. Ευχαριστώ πολύ. Η Νομική Επιτροπή στη συνεδρίασή της 13 Ιουλίου ε, την, ε, ε, ήλεγξε την εντολή του κυρίου Έντουαρτ Σέτσακα και θεωρεί ότι πρέπει να θεωρεί επικυρωθέν με ισχύ από 11 Ιουνίου